Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε νωρίς, γιατί πολύ γρήγορα θα πρέπει να αποχωρήσω για την επανεκκίνηση του Εράσμους Plus με την κυρία Βασιλείου και τον κύριο Μπορίτιο της, από τη Λιθουανία και ο συνάδελφος μετά θα με αντικαταστήσει. Έχετε την ημερήσια διάταξη, υπάρχουν παρατηρήσει προβλήματα. Μια μικρή αλλαγή. Ο κύριος Φίσας θα ήθελε να γίνει η συζήτηση της εκθεσής του αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Στα πρακτικά έχετε τίποτα να το επισημάνετε σας παρακαλώ μέχρι το τέλος της συνεδρίας σας. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Κάποιες γλώσσες δεν καλύπτονται από τη διερμηνία. Δεν ξέρω αν είναι πολλές. Αρκετές μάλλον. Ας μην τις απαριθμίσω, όμως θα το καταλάβετε μόνοι σας όταν δείτε ότι δεν έχετε τη ε, διερμηνία στη γλώσσα σας. Πολωνικά βλέπω, και όλοι οι υπόλοιποι τέλο πάντων ό,τι βλέπετε αναλόγω τη γλώσσα σα. Για το χθεσινό τριμερή διάλογο. Για το θέμα τη ε, ε, πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Θα ενημερωθείτε βέβαια γραπτά. Θα σα παρακαλούσα όμω να μου δώσετε την προσοχή σα γιατί είναι σημαντικά αυτά που έχω να πω. Τριμερής διάλογος λοιπόν για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης συμφωνήσαμε σε ένα θέμα, πλην ενός. Το ποιο ορίζει την πολιτιστική πρωτεύουσα. Το Συμβούλιο επιμένει ότι είναι δική του αρμοδιότητα. Εμείς λέμε ότι είναι εκτελεστική πράξη και ως εκ τούτου είναι θέμα επιτροπής, ούτε καν κοινοβουλίου. Δεν κατέστη εχθές δυνατόν να ακούσουμε διαφορετική τοποθέτηση από την, από την Λετωνία, από την Προεδρία από τη Λιθουανία, από την Προεδρία, ε, είπαν ας πάμε μέχρι πρώτη ανάγνωση. Γελίο μου φαίνεται εμένα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα, μια φορευτική επιτροπή υψηλού επίπεδου η οποία επιλέγει μια πόλη, την προτείνει στην επιτροπή και μετά η επιτροπή την ε, διαβιβάζει στο συμβούλιο για να την επικυρώσει. Εγώ είπα ότι είναι γελίο όταν ούτω ή άλλω μία μόνο πρόταση υπάρχει και μόνο επ' αυτή προτάσεω μπορεί να αποφανθεί το Συμβούλιο, δεν μπορεί να κάνει δηλαδή άλλη πρόταση για πόλη, να γίνεται ε, τόση φασαρία για να ε, αποφασίσει, για να έχει την αρμοδιότητα το Συμβούλιο. Εν περιπτώσει. Έτσι πάμε. Πρώτη ανάγνωση, εάν δεν κλείσει το θέμα μέσα στι 14 μέρε. Και έτσι καθυστερεί λίγο το θέμα, αλλά αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι, α την αναλάβουν. Τώρα, στο σημείο 4 στην δάταξη, έχουμε α, την εκλογή νέου τρίτου, τρίτου αντιπροέδρου που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα αγαπητό Λόταρ Μπίσκι. Έχουμε πρόταση από την ΚΟΕ, την κυρία Ματίνε Μίχελς, τακτικό μέλος πλέον της Επιτροπής μας, προτείνεται ως αντικαταστάτρια του εκλειπώντος. Κυρία Μίχελς, αν θέλετε να σηκωθείτε να σας δουν οι συνάδελφοι. Η νέα σας συνάδελφος είναι εδώ, η κυρία Μίτσελς σας την συνιστώ και θα αντικαταστήσω ως τρίτη αντιπρόεδρο τον κύριο Μπίσκι εάν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή άλλες υποψηφιότητες. Παρακαλώ λοιπόν αφού είναι έτσι να, την, ε, να εγκρίνουμε την εκλογή αυτή. Παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να έρθετε εδώ στη στον αντιπρόεδρο. Και τώρα... Ψηφοφορίες. Εθελοντισμός και εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Έχεις τίποτα, Μάρκο? Όχι, όλα είναι σαφή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρουσίασαν παρατηρήσεις και τροπολογίες. Είναι αρκετά ήρεμος ο κατάσταση ψηφοφορίας. Δεν νομίζω να υπάρχουν ιδιαίτερα πράγματα να προσθέσουμε. Ευχαριστώ εσάς. Ξεκινάμε την ψηφοφορία.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 Η κυρία Κώστα θέλει επαλήθευση της 27. η ψηφοφορία για την 26. 27. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. 15 κατά. 5 υπέρ. Απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη το ίδιο είναι ταυτόσιμο 39 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 40 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε τμήματα η 56 πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 58 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 63, 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 68 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 69 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία δεύτερο τμήμα της 74 Check. Um, the vote is closed. Πέρασε. 13 υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές 82 νομίζω. απερίφθη 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 86 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 87 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές Πολυθεύμα παρακαλώ άρχεται ψηφορία. ψηφοφορία 94 πέρας 12 υπέρ 12, 10 ε, κατά εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100-101 υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απε, ε, ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 15 κατά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 αποχές απερίφθη. Η πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέρα στις μερικές ψηφοφορίες ψηφίζουμε στο σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 22 ψήφισαν, 20 υπέρ, κανένας κατά. Συγχαρητήρια Μάρκο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεργασία στην έκθεση αυτή και τους καλώ βέβαια να υποστηρίξουν αυτή την έκθεση με την ψηφοφορία. Καλώς λέει πρόεδρος, ψηφίζουμε σημείο 5, ε, τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά Αποχές. Επαναλαμβάνουμε. 24 πέρα. Κατά. Επαναληφθεύουμε ηλεκτρονικά. 24. Πέρασε Δέκα υπέρ, έντεκα κατά. Απερίφθη. 26 υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη. 27 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. 17 κατά. 4 υπέρ. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Λίγη γυμναστική το πρωί με την ανάταση τη χειρό θα σα βοηθούσε. Καλώ εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. Αχ, συγγνώμη. Απερίφθη. Και πάμε στο 7. Προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να κάνουμε τις ε, λοιπές ψηφοφορίες όλες μαζί, μπορούμε, τις επόμενες τρεις. Έχετε καμία αντίρρηση. Καλά, εντάξει, 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά αποχές. Ε, πάλι θα έχουμε άλλη ψηφοφορία. What is closed? Άρχεται πέρα ψηφοφορίας, 13 υπέρ, 9 κατά εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και παρακαλώ τις υπόλοιπες τροπολογίες μπορούμε να πούμε ότι τις ψηφίζουμε όλες μαζί είναι τόσο μεγάλες διαφορές 34 μέχρι 45 34 έως 45 όχι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 πέρας προφορίας, 12 κατά 10 υπέρ, απερίφθη, 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ, κατά αποχές επαληθεύουμε, άρχιτε ψηφοφορία για την 16. Πέρας. 13 υπέρ 9 κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Είμαστε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Τελική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονικά. πέρας 22 υπέρ. Καμία ψήφος κατά και συγχαρητήρια αγαπητέ Ζολτάν Μπάγκο. Τώρα αναγκαζόμαι να αποχωρήσω. Θα αναλάβει ο κύριος Φοντάνα την Προεδρία. Oh, Bene, proseguiamo con la... Συνεχίζουμε. E, e, Όπως είπαμε και στην αρχή της συνεδρίασης, πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας ε, διάταξης. Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ε, πτυχές. Οπωσδήποτε ανθρωπολόγος θα επιβεβαίωνε ότι οι τρόποι με τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων προετοιμάζει και καταναλώνει αυτή την τροφή του αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού. Τους. Η Ευρώπη έχει μεγάλο φάσμα γαστρονομικών παραδόσεων και είναι στο επίκεντρο της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η επίγνωση αυτής της κληρονομιάς είναι κάτι σημαντικό. Είναι και στο θέμα του τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού σημαντικό και θα πρέπει να προωθηθεί κυρίως ε, οι νέοι πρέπει να έχουν καλύτερη επίγνωση των κοινωνικών, πολιτισμικών, ιστορικών πτυχών της γαστρονομικής κληρονομιάς της χώρας τους. Αποφασίσαμε λοιπόν να επεξεργαστούμε αυτό το σχέδιο εκθέσεως πρωτοβουλίας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ο συνάδελφος, ο κύριος Φίσας, είναι συγητής μας και θα εκφράσει τις πρώτες του θέσεις του ζητώ να πάρει το λόγο, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υποβληθεί το σχέδιο εκθέσεως της 27 Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο κύριος Φίσας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πιστεύω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θεώρησαν ότι ίσως είναι λίγο περίεργο το θέμα Ίσως να ξεγελάει κάπως ο τίτλος, διότι είναι σημαντικό το θέμα και η διατροφή και η εκπαίδευση στο θέμα αυτό στην ε, Ευρώπη στα σχολεία είναι σημαντικό. Αυτό είναι και η καρδιά του θέματος που συζητάμε. Α, λοιπόν, η αστρονομία εντο... αποτελεί από διάφορες πτυχές της διατροφής. Οι πυλώνες η υγεία, οι συνήθειες διατροφικές και ευχαρίστηση από τη διατροφή. Η διατροφή και η γαστρονομία αφορούν επίσης και κοινωνικές θέσεις, οικογενειακές σχέσεις όλος ιδιαίτερος με τις διάφορες λεπτομέρειες, πολιτισμικές συνήθειες με άλλα λόγια. οικονομική σημασία έχει αυτός το τομέα για την απασχόληση. Έχει και αντίκτυπο και στον τουρισμό η γαστρονομική κληρονομιά και η γαστρονομία αυτή κάθε αυτή αφορά και την ευχαρίστηση να κάθεται κανείς στο τραπέζι και να τρώει. Όταν μιλάμε λοιπόν για γαστρονομία αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις πτυχές που έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στην ποιότητα διαβίωσης των ατόμων. Δεύτερον, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, έχει λέει ότι ένα εκατομμύριο, 200 εκατομμύρια άτομα έχουν πρόβλημα παχυσαρκίας. Και υποφέρουν πολλά από τα, και αντίστοιχα πάρα πολλά άτομα βέβαια υποφέρουν από ε, έλλειψη, από κακή διατροφή στον κόσμο. Εάν συνεχίσουμε έτσι το 2040 ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, θα είναι όλος παχύσαρκος. Ε, λοιπόν, ένα επίπεδο πριν από την υπερβολική παχύσαρκία θα είναι υπέρβαρη. Λοιπόν, η κατανάλωση η παχυσαρκία στα παιδιά βρήκαν στην Αμερική ίσως οδηγήσει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας θα μπορεί τελικά τα παιδιά να ζουν λιγότερο από ό,τι οι γονείς. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Η, παγκόσμια, οργάνωση της ε, εργασίας και της οικογενικής ζωής ε, οδηγεί σε αυτό διότι μαγειρεύουν πολύ πιο βιαστικά στο σπίτι. Ε, η ζωή γίνεται καθιστική περισσότερο στο σπίτι, αδρανής και τα παιδιά ε, μετακινούνται όλο και λιγότερο με τα πόδια για να πάνε στο σχολείο, παίζουν λιγότερο στα πάρκα και στους δρόμους. Και για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό. Ε, και ε, κάθονται περισσότερο και στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο, παίζουν με τις παιγνιδομηχανές. Περισσότερο καθιστική ζωή ζουν τα παιδιά. Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν καλύτερα στα παιδιά, στα σχολεία, τη σημασία που έχει φυσική άσκηση και σωστή διατροφή και γαστρονομία. Θα πρέπει λοιπόν να παίξει αυτό το ρόλο το σχολείο. Λοιπόν, 10 ευρωπαϊκές χώρες, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, μεταξύ αυτών και η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό τη σωστή διατροφή μαζί και η Σουηδία. Ελπίζουμε και άλλε χώρε επίση να θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο που δημιουργήθηκε σωστή διατροφή στην Ευρώπη. Πρέπει να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων χωρών. Και λοιπόν με κάποιε συνεδριάσει του φορέα αυτού έγινε μεγάλη συνεδρίαση στη Μαδρίτη το 2010 και επικεντρώθηκε επί δύο βασικών θεμάτων. Η διατροφή στο σχολικό πρόγραμμα και η ρύθμιση του θέματος των διαφόρων ποτών και των τροφών που δίδονται στα σχολεία. Θα πρέπει λοιπόν να προτρέχουμε τη διατροφή που σχετίζεται με την παιδεία αλλά και διάφορες πολιτιστικές και οικονομικές πτυχές της γαστρονομίας να μην λησμονούμε ότι η UNESCO καθορίζει την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, όλη την κληρονομιά που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και αποτελείται από την γνώση των διαφόρων εθήμων, ηθών, τεχνικών που διαβιβάζονται από γενιά σε γενιά και που δίνουν στην κοινότητα και στην ομάδα ένα συνέστημα ταυτότητας και συνέχεια συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόθεση του σεβασμού της πολιτισμικής ποικιλομορφία και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Γι' αυτό το 2010 η UNESCO συμπεριέλαβε στον κατάλογο τον αντιπροσωπευτικό του της πολιτισμικής κληρονομιάς της ανθρωπότητα, ανθρωπότητας, τη μεσογειακή δίαιτα Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Ελλάδα, και τη διατροφή και στη Γαλλία και παραδοσιακή κουζίνα ε, και του Μεξικού. Παραδοσιακή κουζίνα του Μεξικού. Ε, ε, λοιπόν, πάνω σε αυτά τα στοιχεία που ανέφερα ο βασίζεται η έκθεσή μου, αν και δεν φαίνεται πρώτη ματιά, μπορεί αυτό το θέμα να έχει μεγάλο αντίκτυπο εις μελλοντικέ γενιέ για το μέλλον των παιδιών μα. Ευχαριστώ Πρόεδρο, βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα. στη διάθεση των συναδέλφων, αν υπάρχουν κάποιε ερωτήσει ή κάποιε παρατηρήσει για το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φίσας, το λόγο. Ε, κυρία Μακλάρκιν έχει τώρα. Ευχαριστώ. Πράγματι χαίρομαι που επιτέλους ε, συζητάμε την ε, γαστρονομική κληρονομιά. Είναι μια έκθεση που εγώ πρότεινα εδώ και κάποια χρόνια και χαίρομαι ως ιδιαίτερος που τελικά εμφανίζεται. Η γαστρονομία είναι το κεντρικό σημείο και θα πρέπει να εξετάσουμε εκ του και στην χρήση της λέξης γαστρονομία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην μπαίνουμε σε περιοχές που είναι εκτός ε, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ε, της Πολιτιστικής. Ε, η, διατροφική, η διατροφή είναι πολύ σημαντική, αλλά η υγεία δεν είναι θέμα της Επιτροπής. Μπορούμε να το αναφέρουμε στα θέμα την υγεία, αλλά δεν θα πρέπει να εστιάζεται έκθεση πάνω στην υγεία. Θα ήθελα η έκθεση αυτή να γιορτάζει, να περισσότερο να τονίζει τις διάφορες πολιτισμικές κληρονομιές στην γαστρονομία και να χαιρετήσουμε και να απολαύσουμε και να γιορτάσουμε για όλες τις, τις τροφές που έχουμε στις διάφορες περιοχές. Είναι ποικιλομορφία που προέρχεται από τα διάφορα είδη τροφίμων που παράγουμε και τη διατροφή μας και είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν στις πολιτισμικές πτυχές και να δούμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις διάφορες τεχνικές μαγειρέματος και αυτό έχει αξία σαν παιδεία, αλλά πρέπει να φυλάξουμε την κληρονομιά ε, να καταλάβουμε πώς έχει αναπτυχθεί η γαστρονομική κληρονομία επί σειρά ετών. Ε, είναι, με ενθουσιάζει. Εγώ τα Ανατολικά Μίτλαντ εκπροσωπώ, εστιαζόμαστε πολύ στη διατροφή και τα ντόπια προϊόντα που παράγουμε στα αστικά. Έχουμε περίφημο λουκάνικο, ε, το, το λουκάνικο του Lincolnshire και έχουμε το τυρί Στίλτον και την πίτα, την pork pie και με χοιρινό. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ. Ε, ο τουρισμό, το εμπόριο, υπάρχουν διάφορε πτυχέ λοιπόν. Λοιπόν, ε, ελπίζω να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση ούτω ώστε να το τονίσουμε, να το γιορτάσουμε, να μην θεωρήσουμε ότι είναι ελαφρύ θέμα. Δεν είναι ελαφρύ, είναι ένα κομμάτι τη αυτοτητά μα τη κληρονομιά. Οι Ιταλοί είναι υπερήφανοι, απίστευτα υπερήφανοι για τη δική τους γαστρονομική κληρονομιά, οπότε και εμείς στη Βρετανία είμαστε. Um, θα ήθελα να εστιαστώ σε μια άλλη πτυχή αυτού. Ο συνδυασμό τη εκτίμηση δύο διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, αυτό είναι ένα άλλο τομέα ο οποίο αντικατοπτρίζεται στην περιοχή μου. Εκεί έχουμε μεγάλο ασιατικό πληθυσμό που έχει έρθει και έχουμε αναπτύξει πραγματικά συγχώνευση κουζίνας, αγγλοϊνδική γαστρονομική κληρονομιά έχουμε γαστρονομικό ταξίδι θα έλεγα και έτσι έχουμε αναπτύξει αυτή την κληρονομιά και αυτό ε, το εκτιμούν και έτσι εντάσσεται περισσότερο κόσμο στην κοινωνία και καταλαβαίνουμε ημέν τους δε καλύτερα. αφού θέλουμε να τονίσουμε τα προϊόντα της χώρας μας και αυτό που είναι βρετανικά στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσουμε τη γαστρονομία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στον άλλο καλύτερα. Και αρχίζω και πεινάω, ακόμα και το σκέφτομαι. Έπρεπε να είχα φάει πρωινό σήμερα, το πρωί ξέρα. Αλλά προσβλέπω συνεργασία με τον κύριο Φίσα σε αυτή την έκθεση και τι συζητήσει για τα υπέροχα τρόφιμα, τα υπέροχα φαγητά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Μακλάρκιν. Επόμενη συνάδελφα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κάμερεβερτ. Ευχαριστώ πολύ και την συνάδελφο για την προετοιμασία της εκθέσεως. Ε, η σκιώδη συγκέντρια εκ σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Μου έχει δώσει τις προτάσεις της, θα σας τη διαβάσω, θα προσπαθήσω να σας τα πω με δικά μου λόγια. Η γαστρονομία είναι πολύ σημαντικό συστατικό κομμάτι ε, της κουλτούρας μας, του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και της πολιτισμικής μας πολυμορφίας που τόσο πολύ εκτιμούμε και θέλουμε να προστατέψουμε. Η Ιζαμπέλ Τομάν, λοιπόν, και ο συγκήτρια μου σημείωσε επίσης στα όσα είπε και η κυρία Μακλάρκιν, ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στα χωράφια άλλων ε, επιτροπών αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για γαστριμαρχική πολυμορφία εάν δεν γνωρίζουμε τι είδους τρόφιμα παράγονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο όταν μιλούμε για τοπικά προϊόντα και, την, και θέλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή τοπικών προϊόντων ώστε να μην ε, φτάνουν από το ένα άκρο της Ευρώπης μέχρι το άλλο οι τροφές, χρειάζεται η ενίσχυση και του τομέα της γεωργίας και της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ιζαμπέλ Τωμά, αναφέρθηκε άλλωστε και από τον Σαντιάγο αλλά και από άλλους, ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ε, κατάρτισης και της μετεκπαίδευσης. Ε, φυσικά και χρειάζεται να έχουμε πολύ καλό προσωπικό στο χώρο της γαστριμαργίας ε, και στην κουζίνα και στην εξυπηρέτηση στην αίθουσα, αλλά και ε, ανθρώπους ικανούς που θα γνωρίζουν τι αγοράζουν, ποια είναι τα ποιοτικά προϊόντα. Αλλά επίσης θέλουμε και μία προοπτική για το μέλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Και πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας να καταρτίζονται, να ε, εκπαιδεύονται, να μαθαίνουν τα ίδια να μαγειρεύουν καταρχάς. Εγώ στο σχολείο δεν είχα αυτή την ευκαιρία, παραδείγματι, πώς ε, χρησιμοποιούμε τα συστατικά, ε, πώς τα βάζουμε μαζί σε μια κατσαρόλα για να φτιάξουμε ένα νόστιμο φαγητό και επιπλέον αυτού πιο εξειδικευμένα δυνατότητες εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης για τους τόσους μάγειρους στην Ευρώπη που μπορούν να μάθουν ο ένας ε, για την κουζίνα του άλλου, επί παραδείγματι. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο ε, κέρδος, πιστεύω, και εγγύηση για το μέλλον. Η έκθεση προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία, πιστεύω, το θέμα αυτό να το ε, καλύψουμε και σε σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες γενικά, αλλά και στα επιμέρους σημεία του. Με, όπως και η Ιζαμπέλ πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση και μπορούμε να έχουμε στο τέλος μετά την ψηφοφορία μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Σκούρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση που θελήσαμε πολύ να υλοποιηθεί, όπως έλεγε και η συνάδελφος Μακλάρκεν. Θέλαμε και από πλευρά της ομάδας τους να μιλήσει αυτό το θέμα είναι ένα ζήτημα που γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Γιατί έχει πάρα πολλέ ε, συνέπειε. Υπενθυμίστηκε ότι πρέπει να παραμείνουμε εντός των αρμοδιοτήτων μας, να μην μπούμε σε αρμοδιότητε άλλων των επιτροπών. Προφανώς όμως το θέμα απαιτεί εξέταση πολλών πτυχών. Η πολιτισμική πτυχή ήδη υπενθυμίστηκε από τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό. διότι είναι κάτι πασίγνωστο στην Επιτροπή. Είναι μεγάλη κληρονομιά ποικιλομορφίας και πλούτου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και πτυχές εκπαιδευτικές. Γιατί το λέω αυτό. Διότι πιστεύω ότι στις κοινωνίες μας είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διδάξουμε να επεξεργαζόμαστε τα ε, να μάθουμε και να τρώμε. Πολλοί κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και γιατροί μας λένε ότι τρώνε άσχημα τα, οι ανήλικοι τα παιδιά. Έχουν κακή σχέση με τη γαστρονομία, τα τρόφιμα και την ε, κουζίνα. Αυτή η πτυχή, χωρίς να μπούμε σε αρμοδιότητες που δεν είναι δικές μας, πρέπει να εξεταστούν κατά κάποιο τρόπο στην έκθεση αυτή. Διότι σήμερα πολλά από τα προβλήματα των νέων, έχουμε και αυτή την αρμοδιότητα βλέπετε σε αυτή την Επιτροπή, αφορούν και τη σχέση των παιδιών με τα τρόφιμα και πώς τα χρησιμοποιούν. Παρόλο που αναφέρθηκαν διάφορα θέματα για την βουλημία, την ε, παχυσαρχία κλπ. και την ανορεξία. Πολλοί νέοι τρώνε με τρόπο αρνητικό γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Διότι Θέλουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ταυτόχρονα να εξετάσουμε και το θέμα τη αστυνομία που είναι μια κληρονομιά τη Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Σκούρια. Μήπω κάποιο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο, κάποιο εκπρόσωπο. Θέλει κανεί το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Ορίστε, παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω το όνομά σα. Αν μπορούσατε να συστηθείτε. Φίλιξ Ρόν το όνομά μου και δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ήρθα για να σας ε, εξηγήσω εν συντομία το τι έχει προσφέρει το πρόγραμμα Λεωνάρτο Νταβίντσι, αυτό που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση στο παρελθόν, και τώρα το νέο Erasmus+. τα οποία θα κάλυπτε αυτά τα θέματα που συστήθηκαν τώρα. Ε, έριξα και μια ματιά στην τράπεζα δεδομένων μας για να δω, έχω μια επισκόπηση των ε, ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπάρχουν. Είτε πρόκειται για ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ε, εστίασης. Έχουμε τα τελευταία χρόνια ολοκληρώσει 300 προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν ε, προσφέρει και δυνατότητα στην κινητικότητα, δηλαδή πρακτική εξάσκηση από το ένα κράτος στο άλλο και έχουν χρηματοδοτήσει αυτές τις πρακτικές εξασκήσεις, είτε, έχουμε, είτε έχουν χρηματοδοτήσει ή διευκολύνει συνεργασία μεταξύ ειδικών σχολών κατάρτισης, τόσο για ε, υποστήριξη των μαθητών σπουδαστών όσο και για ανταλλαγή τεχνολογίας κατάρτισης και άλλα. Και θα ήθελα για να δώσω κάποια παραδείγματα να απαντήσω τα εξής. Λέγεται ότι πρέπει να διαφυλαχθεί. Βεβαίως πρέπει να διαφυλαχθεί. Αυτό που υπάρχει όμως και μπορεί να διαφυλαχθεί κάτι και στο σπίτι του καθενός αλλά και ακόμα στο εξωτερικό. Επί στην σαχαροπλαστική. Η ε, Σόφια, στη Σοφία με ε, ένα σχολείο ειδικό ε, το οποίο μπόρεσε να αποστείλει στο Βέλγιο, τις Βρυξέλλες, συγκεκριμένα την Αμβέρσα και τη Βρύγη, φοιτητέ του, οι οποίοι ήρθαν και έμαθαν πώς γίνεται εδώ, στο Βέλγιο, η ζαχαροπλαστική και κυρίως ποια είναι η τεχνική για την λεγόμενη βελγική πραλίνα, τα σοκολατάκια τα βελγικά και βέβαια αυτή την τεχνογνωσία την πήραν μαζί τους επιστρέφοντας στη Βουλγαρία. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Επίσκεψη και πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό. Άλλο, ε, από επαγγελματικέ σχολές πάλι, παράδειγμα, μία ένωση δημοσίου συμφέροντος, ε, όπως ονομάζεται, για την συνεχή και διαβίου μάθηση στην Κάτω Νορμανδία και είχαμε ένα Land College ε, ανώτερης εκπαίδευσης από τη Σκοτία το οποίο επισκέφθη ε, την σχολή και μάλλον μαζί με την, και με τη σχολή των ξενοδοχειακών ε, υπηρεσιών του Καλβαντός και αντίστοιχα μια σχολή για ε, υπηρεσίες ξενοδοχειακές της Γερμανίας και άλλη μία της ε, Πολωνίας από το Λότσι ε, έγινε μια συνεργασία μεταξύ αυτών των σχολών. Ο στόχος ήταν ο εξής, οι σπουδαστές της σχολές αυτές να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν, να γνωρίσουν ξένα τα μενού ή τον τρόπο διατροφής από άλλες χώρες να δούνε λοιπόν τα μενού κάποιες άλλες χώρες, ε, τα πιάτα μιας άλλης χώρας, να μάθουν πώς παρασκευάζονται αυτά. Πολύ ενδιαφέρον ε, ήταν και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο λεξιλόγιο, στη γλώσσα δηλαδή της χώρας από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο πιάτο, άρα υπήρχε μια βασική γλωσσική μάθηση και βέβαια άλλες πτυχές ε, πρακτικές για το πώς δουλεύουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, πώς συγκεκριμένα παρασκευάζουν ε, το πιάτο, όχι μόνο δηλαδή ανταλλαγή συνταγών. Και επίσης ε, συνεχίστηκε ο στόχος δεν ήταν μόνο μια συνεργασία διαδικτυακή βέβαια, αλλά η δυνατότητα οι φοιτητέ σπουδαστέ αυτών των επαγγελματικών σχολών να προετοιμάζονται εγκαίρως μέσω της διαδικτυακής αυτής προσπάθειας και της σελίδας που ε, κατασκευάστηκε να προετοιμάζονται εγκαίρως λοιπόν για, ένα, για μια πρακτική εξάρεσκηση στο εξωτερικό. Με το Erasmus Plus συν θα έχουμε αντίστοιχες δυνατότητες ε, για ανταλλαγές ε, επισκέψεων και για τις επαγγελματικές σχολές, δυνατότητες που είχαμε και στο παρελθόν βεβαίως και για, τις, ε, ε, για τη σχολική μάθηση και στον τομέα που αναφέρεται ε, για την προσέγγιση του, της διατροφικής και της μαγειρικής μέσα από το σχολείο θα μπορούσε το ε, κοινό σχολείο, το κανονικό σχολείο να καλύψει αυτό, αλλά επίσης θα μπορούσε και μεταβατικά να υπάρξουν συνεργασίες με επαγγελματικές σχολές. Αυτό είναι μια δυνατότητα που προσφέρει το Erasmus 2+. Ε, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Θα δώσουμε ξανά το λόγο στον κύριο Φίσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα υπόθηκαν Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους και ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να πω στην κυρία Μακλάρκεν ότι χαίρομαι ιδιαίτερο που είναι σκιώδης ε, εισηγήτρια για την έκθεση αυτή της, ε, την ομάδα της. Και εγώ ε, ήθελα να συμπεριλαμβάνω δύο πυλώνες στην έκθεση. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, την παιδεία στα σχολεία, ένας πυλώνας. Δεύτερο όμως πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν να τονίσουμε την πολιτισμική κληρονομιά μας από γαστρονομική πλευρά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για να εντάξουμε, το να εντάσσουμε άλλες, άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες μέσω της γαστρονομία. Πάντα θεωρούσα ότι η γαστρονομία είναι σημαντικό κομμάτι πολιτισμικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το τομέα. Η ιδέα μετά που αναφέρθηκε του να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντική, Πέτρα. Τα παιδιά μαθαίνουν τους γονείς τους καμιά φορά πράγματα. Παραδείγματος χάρη για τα απόβλητα ε, στη γενιά μου τα πετάγαμε παντού. Σήμερα τα παιδιά λένε όχι. Αυτό το βάζει στην πράσινη σακούλα, το άλλο το βάζει στη γαλάζια σακούλα κλπ. Τα παιδιά διδάσκουν του γονεί πώ να ξεχωρίζουν τα διάφορα ε, σκουπίδια. Αν δίνουμε αυτέ τι αρχέ στα παιδιά μα στο σχολείο για το πώ μπορούν να τρέφονται καλύτερα, ούτω ώστε τα παιδιά να παίρνουν τι αποφάσει, ε, αυτό είναι σωστό, θα είναι καλό. Μπορεί να γίνει και μέσω τη οικογένεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ρόλο των σχολείων. Και μετά είναι και το θέμα της ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα. Όταν συζητάμε την ε, κρίση στην Ευρώπη, η επαγγελματική κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική και οι οικονομικές πτυχές και η ιδέα του να βρίσκει κανείς δουλειά μέσω της γαστρονομίας ίσως θα πρέπει να μην μείνει στο περιθώριο σαν ιδέα, είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα. Και θα το συμπεριλάβουμε αυτό στην ε, έκθεση. Μάρκο, αναφέρθηκες στις κακές συνήθειες που υπάρχουν όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή και πόσο επικίνδυνα είναι αυτά για την υγεία. Ναι, θέλουμε να το καλύψουμε αυτό, το θέμα της βουλημίας και της ανορεξίας. δεν είναι μόνο προβλήματα των νέων, αλλά είναι κυρίως των νέων. Και είμαστε υπεύθυνοι για ζητήματα πολιτικής που αφορούν τους νέους. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικές ασθένειες των νέων και πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Μετά, σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγματι υπήρξαν κάποια προγράμματα από το Λεωνάρντο και χαίρομαι που ακούω ότι θα συνεχιστούν και ότι δεν θα εξαφανιστούν όπως είχαμε ακούσει στην αρχή και το Erasmus Plus σε συνδυασμό με την επαγγελματική κατάρτιση και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και των καλύτερων ευρωπαϊκών συνταγών, πράγματο χάρη, πώ μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα προϊόντα. Όλα αυτά διδάσκονται στα σχολεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που άκουσα από η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει συντονιστεί στο ίδιο μήκο κύματο. Και βιάζομαι να ξεκινήσω δουλειά πάνω στο θέμα αυτό και να συνεργαστώ με του κοιόδη συζητητέ, την κυρία Μακλάρκιν τον Τόμα δεν ξέρω από του από την ΚΟΕ, αν ήδη έχουν καθορίσει σκιώδεις συγητές από τι ομάδε του, Ελπίζω να καταλήξουμε σε, στην ευρύτερη δυνατή συνένεση πάνω αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι νομίζουν κάποιοι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Φίσα. Εγώ τώρα θα έλεγα να πάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης προετοιμασία για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο οπτικοκουστικός τομέας αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα. Υπάρχει αυξανόμενη σύγκληση στον οπτικοκουστικό τομέα με την ανάπτυξη διαφόρων υβριδικών μηχανισμών όπως είναι οι διάφορες τηλεοράσεις ευφυής που συνδέονται με το διαδίκτυο. Όλα αυτά δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες για την παροχή υπηρεσιών και συν και χάνονται τελικά τα διάφορα σύνορα μεταξύ καταναλωτών, τηλεόρασης και διαδικτύου. Λοιπόν, ανακατανάλωση των τικοστικών προϊόντων σημαίνει ότι του καταναλωτή μια ευρύτερη ε, ε, πρόσβαση σε ευρύτερο περιεχόμενο, αλλά είναι και μια πρόκληση που αφορά τον ανταγωνισμό ή τα πνευματικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υιοθέτησε μια πράσινη βίβλο όσον αφορά την προετοιμασία ενός οπτικοακουστικού ε, τομέα να υπάρξει πλήρη σύγκληση στον, στον τομέα και η Επιτροπή μας θεώρησε ότι έπρεπε να ετοιμάσουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλής ε, και η συγγήτριά μας είναι η κυρία Βεραίν, η οποία θα εκφράσει τις πρώτες σκέψεις στο θέμα. Το σχέδιο εκθέσεως πιθανότατα θα υποβληθεί στις 27 ε, Νοεμβρίου. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, στις 24 Απριλίου κατέθεσε την πράσινη βίβλο, της προτάσεις δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ε, ξεκίνησε η συζήτηση για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο. Εμείς κάναμε μια έκθεση για τις ε, ευφυείς τηλεόρες, τηλεοράσεις, τα ευρυδικά αυτά, τις ευρυδικές αυτές συσκευές, συνδεδεμένες ε, και με αυτή την πρόταση και την επιτροπή, ξεκινάει η συζήτηση για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο. Η πράσινη βίβλος λοιπόν ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην ε, παραγωγικότητα για το μέλλον αποτελεσμάτων από την οδηγία για τα οπτικοακουστικά, τις αλλαγές υποδομές, τρόπους χρηματοδότησης, μοντέλα χρηματοδότησης, ε, ιδιαιτερότητες, τα οπτικοακουστικά, ψηφιοποίηση στον όλο τομέα και ιδιαίτερα σημαντικό είναι να δούμε τι είδους αλλαγές μπορεί να προκύψουν ως προς την χρήση των συχνοτήτων. Τι είδους φάσμα χρειαζόμαστε, εάν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο φάσμα από ό,τι παραδοσιακά προτινόταν για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση, αλλά βέβαια υπάρχει άλλη έκθεση που ασχολείται με το θέμα αυτό εντατικά. Στην πράσινη βίβλο ε, γίνονται και προτάσεις για την ε, αγορά, ε, κατακόρυφη αλλά και οριζόντια ολοκλήρωση του τομέα, ενσωμάτωση του τομέα. Η κατακόρυφη είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε να κάνουμε με τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες και η, την εικόνα αυτού του πεδίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βέβαια παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, σε μεγάλο βαθμό, ε, σε περιορισμένο βαθμό πλέον αρμοδιότητα της Ευρώπης, μόνο μια προσπάθεια για κοινή ανάπτυξη των μέσων ε, μπορούν να επιχειρήσουν τα κράτη-μέλη και καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα. Κύρια προβλήματα λοιπόν, αν προκειμένου είναι η σύγκληση, δηλαδή η παράλληλη ανάπτυξη των, των υπηρεσιών των μαζικής ενημέρωσης κατά τρόπο που μέχρι τώρα ήταν πολύ διαφορετική να προχωρούν εκ παραλλήλου και με μειωθό τρόπο, γραμμική μη γραμμική. Μετά έχουμε νέους παρόχους υπηρεσιών από το χώρο των τηλεπικοινωνιών αλλά και παρόχους υπηρεσιών ε, over the top όπως ονομάζονται οι οποίοι δεν παρακολουθούν τις παραδοσιακές σαφείς δομές που υπήρχαν στους τομείς αυτούς και έτσι μπορούν να διαταράξουν σημαντικά την αγορά. Ως προς την ψηφιοποίηση των, της τεχνολογίας εκπομπών και τα υβριδικές συσκευές έχουμε και τις παραδοσιακές βέβαια νομοθεσίες που ίσχυαν ε, για τους τομείς εκτός ίντερνετ, δηλαδή για τις εκπομπές με ραδιοκύματα, αλλά και νέα νομοθετήματα που αφορούν το ίντερνετ. Ε, σε σχέση με τον καταναλωτή, την νεολαία, την προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων και, τις, ε, και το από το μέσα μαζικής ενημέρωση υπάρχει σχετική οδηγία. Ε, Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η προστασία της ποικιλομορφία και του χαρακτήρα του πολιτιστικού προϊόντος ως ε, αγαφού ιδιαίτερα σημαντικού για τις κοινωνίες στην Ευρώπη. Επιπλέον έχουμε ερωτηματικά. Χαίρομαι για την ε, διεύρυνση της ε, μονοδιάστατης συζήτησης για το τηλεοπτικό κόσμο έτσι ώστε να ανοίξει το πεδίο και πάλι εδώ η κατακόρυφη ολοκλήρωση θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Προκύπτουν βέβαια νέες ε, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τους εμπλεκόμενους στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξυγκλίνουν στις αγορές λοιπόν τι θα μπορούσε να είναι. Όταν ε, κατά πρώτο λόγο έχουμε είτε τηλεόραση είτε την παραδοσιακή ε, μορφή εκπομπής που πια θεωρούνται οι δεινόσαυροι των μαζικής ενημέρωσης και υποχωρούν και μεγάλο μέρος ε, των καταναλωτών ε, πλέον, μερίδιο μάλλον των καταναλωτών παραμένει ακόμη πιστό στην παραδοσιακή μορφή εκπομπής αλλά τίνει όλο και περισσότερο να αξιοποιεί τα κινητά, τις κινητές συσκευές. Το ζήτημα το περίφημο σύστημα του, streaming, ότι ένας νεαρός μπορεί να έχει στα χέρια του ένα iPhone, ένα τηλέφωνο FES, να έχει και ένα κομπιούτερ παραδίπλα και να παίζει και η τηλεόραση λίγο πιο μακριά και να παρακολουθεί ταυτόχρονα διαφορετικές ε, εκπομπές. Παράδειγμα ε, που ακούστηκε, μια μάνα που μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού της, παίζει τηλεόραση, είναι και το κομπιούτερ αναμένο και παίζει ο μικρός με το κομπιούτερ και από την άλλη με το smartphone ε, επικοινωνεί σε κάποιο chat. Και μπαίνει λοιπόν η μητέρα και βλέπει αυτή τη σκηνή και λέει στο γιο μα τι κάνεις, α δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια μαζική επικοινωνία και ροή, αλλά ε, πρέπει και η αντίληψη να εξεταστεί στην υπόθεση αυτή, η αντίληψη του τι κάνουμε. Λοιπόν, ε, η σύγκληση στον τομέα αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μεγάλη ευκαιρία για κοινοτομία, γιατί θα χρειαστούν νέε μορφέ συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και τομέων. Ε, περιεχόμενα στο τελικό, σε διαφορετικό τελικό ε, αντικείμενο υποδοχή υποδοχέα, σε διαφορετική συσκευή δηλαδή, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά και επίσης θα πρέπει να επαληθευτεί η σκοπιμότητα της εισαγωγής της οδηγίας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εισήχθη αυτή η οδηγία και σε ποιο βαθμό τους στόχους οποίους υποτίθεται εξυπηρετούσε όταν εισήχθη μπορεί να τους εξυπηρετήσει τώρα με τον τωρινό κόσμο και την ψηφιακή εποχή. Και βεβαίως εάν μπορεί ή χρειάζεται να γίνει προσαρμογή των αγορών στις νέες συνθήκες, πρέπει ίσως να γίνει αντιπαραβολή με ισχύουσες νομοθεσίες που έχουν επίδραση στο χώρο των μαζικής ενημέρωση. Παραδείγματι αυτή που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αδειοδότηση μουσικών και άλλων πολιτιστικών έργων, το ζήτημα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, των εκπομπών, ε, ραδιοσυχνοτήτων και των σχετικών συσκευών και βέβαια δεν μπορούμε να λησμονήσουμε από αυτό και το μεγάλο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Ε, όταν γίνει η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού δικαίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία αυτών ως παράγοντα ε, πολιτιστικού, ως προϊόντος πολιτιστικού σε κάθε τομέα, σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς όμως. Η προσβασιμότητα επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι ε, ξέρετε ότι αν κάποιος θέλει να διαθέσει ένα προϊόν και να έχει επιτυχία μέσα από το ίντερνετ, πρέπει να έχει και την ορατότητα και την δυνατότητα πρόσβαση διαφορετικά ε, και αθέμητος ανταγωνισμός ε, και στρέβλωση του ανταγωνισμού αποτελούν σημαντικούς κινδύνους, κυρίως όταν θέλουμε να έχουμε μια πολιτιστική πολυμορφία η ουδετερότητα του δικτύου επίσης. Ε, πιστεύω ότι αυτό θα αποτελούσε μια ε, εγγύηση για, που θα μπορούσε να αποτρέψει τις τρευλώσεις και πρέπει να μπει στους στόχους μας για, έναν, για τις συγκλίνουσες αγορές με τον ορίζοντα 2020, για τις υπηρεσίες 2020, ε, για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ουδετερότητα λοιπόν αυτή, και ιδιαίτερα αν θέλουμε να δώσουμε σε μια υπηρεσία την προτεραιότητα, θα πρέπει να εξετάσουμε αν αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα δεν ε, ε, μειώνεται ή δεν μπαίνει στο περιθώριο μια άλλη μορφή υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ουδετερότητα. Και πρέπει βέβαια αυτό να το συζητήσουμε και να επαληθεύσουμε τους ε, νόμους, την νομοθεσία, τους ορισμούς που ισχύουν και τι είδους προτεραιότητες ακολουθούν σε σχέση με τις δομές, κυρίως στην έννοια της πλατφόρμας. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες αλλά και σε περιεχόμενα υπηρεσίες ε, σε διαφορετικά διαφορετικές συσκευές ή μέσω διαφορετικών συσκευών μπορεί να έχει μια επιχείρηση, δηλαδή η συγκέντρωση αυτής της ε, πυκνότητας πληροφοριών σε ορισμένες επιχειρήσεις είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Ε, οι εφαρμογές επί παραδείγματι, οι οποίες ε, δεν διατίθενται σε σελίδες ή δεν περνούν ε, ε, στο διαδίκτυο γιατί δεν αντιστοιχούν στην ηθική διάσταση της επιχείρησης και αυτό βλέπουμε ότι στις Ρωμανίες πολιτείες έχουν συνέπειες. Στόχος επίσης πρέπει να είναι ή δεν περνούν στο διαδίκτυο γιατί δεν αντιστοιχούν στην ηθική διάσταση της επιχείρησης και αυτό βλέπουμε ότι στις ΗΠΑ σε παραδείγματα έχει συνέπειες. Στόχος επίσης πρέπει να είναι η εξασφάλιση, η προστασία της ε, πολυμορφίας και βέβαια η κατάλληλη χρηματοδότησή της πρέπει να υπάρξει ρυθμιστική ρύθμιση όπου αναγνωριστούν οι σχετικές ανάγκες για έλεγχο, για ε, αντιμετώπιση κινδύνων επιρροής της ε, διαμόρφωσης της κοινή γνώμης. Η πλατφόρμα και ο ορισμός της πλατφόρμας θα πρέπει να ε, αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, πολύ πιο συγκεκριμένα, γιατί ορισμοί υπάρχουν, υπάρχει κανονισμός πλατφόρμας για τα καλωδιακά δίκτυα, τους δορυφόρους, κάποιους τρόπους μεταφοράς της πληροφορίας. Ο ορισμός της πλατφόρμας υπάρχει λοιπόν, αλλά το search neutrality, το λεγόμενο, η λεγόμενη αρχή της ε, ουδετερότητας της αναζήτησης και βέβαια η, η ανάγκη εξυπηρέτηση διαφορετικών τελικών συσκευών ε, δεκτών, ε, θα πρέπει να ληφθούν και αυτές εδώ υπόψη. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση των προτινομένων δια, τάξεων με υφιστάμενα νομοθετήματα που έχουν να κάνουν παραδείγματι με τον ε, των ανταγωνισμό, με τις τρεύρε των αγορών κτλ. Θα πρέπει να επαληθευτεί δηλαδή αν χρειάζονται ή αν ήδη καλύπτονται από κάποια άλλα νομοθετήματα. Αυτό για κάθε τομέα των μέσων μαζική ενημέρωση και ανάλογα με τις ε, ε, με την αντανάκλασή τους. Στόχος θα πρέπει να είναι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάθε τομέα των μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε πρόκειται για παραγωγούς ε, ραδιοεκπομπών, ε, είτε για οτιδήποτε άλλο, να έχουν το, ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ώστε να μην προκύψουν στρεβλώσεις. Η σύγκληση θα πρέπει να, προτείνει ευκαιρίες περισσότερο, και δυνατότητες για ανάπτυξη και νέων ε, προτύπων, νέων μοντέλων επιχειρησιακών και νέων μοντέλων δραστηριοποίησης ε, με διαφορετικές προσφορές και αυτό όχι μόνο με σκέψη, με μέλημα πόσο θα κοστίσει κάτι, αλλά με ουσιαστικό ε, στόχο το αποτέλεσμα της προτινόμενης υπηρεσίας. Θα χρειαστεί ενδεχομένως να αναλάβουν δράση δομές ε, στους διάφορους τομείς ε, και να ανατρέψουν τα εσκεμένα ως προς ε, τα πρότυπα λειτουργίας αγοράς για να εξυπηρετηθούν νέες ανάγκες και πρότυπα κατανάλωσης σε, αυτή, σε αυτό το συμπολιτισματικό τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν. Ε, πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε πρόσδεκτο επακριβώς εντοπίζει τα σημαντικότερα ζητήματα που θα αφορούν τον οπτικοκουστικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Καλή βάση για συζητήσεις που θα λάβουν χώρα. Επανειλημμένα συζητήσαμε τη σημασία του οπτικοκουστικού τομέα. Σημασία στον αφορά ανάπτυξη και θέση απασχόλησης και τι μπορεί να πετύχει για τον δημιουργικό μας τομέα και τον πολιτισμικό. Μετά καινοτομία, ανάπτυξη, ανταγωνισμό, αυτές οι πτυχές εξαρτώνται από την ε, σύγκληση που θα λάβει η χώρα. Αυτό συνεπιφέρει πολλές προκλήσεις, αναφέρονται στο έγγραφο. Χρειάζεται χρόνος για να κατανοήσουμε πώς η τεχνολογία θα αναπτυχθεί, πώς θα συμβούν όλα αυτά. Έτσι θα βρούμε σωστές λύσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του εγγράφου που θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, υποδομές. Χωρίς επαρκή υποδομή η αγορά δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί, δεν θα υπάρξει καινοτομία. Στην κοιμοκλογική περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση ακόμα σε βριζονικές υπηρεσίες. Πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ατζέντα που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να ωφεληθούν από τις ε, εξελίξεις και να έχουν επαφή με το διαδίκτυο και το μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την ΕΦΗ e τηλεόραση συνδέεται με το διαδίκτυο ε, είναι αυτό κάτι που θα προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ληφθεί υπόψη στην Πράσινη Βίβλο. Συζητούμε τον κατακαιρματισμό που υπάρχει, πώς καταλήξαμε εκεί, πώς θα πετύχουμε διαλειτουργικότητα, διασυνοριακή προσέγγιση, Είμαστε στην αρχή της επανάστασης και χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλάβουμε τα προβλήματα πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε λύσεις. Άρα πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας περισσότερο χρόνο να βρούμε σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα ανακύψουν. Για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό πρέπει να επιτρέψουμε το διαδίκτυο να δώσει τη δύναμη που πρέπει στους πολίτες και να μπορούν να βγάλουν άκρη στις πληροφορίες οι άνθρωποι και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που επιθυμούν και να καλύψουν τις προσωπικές ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα διαφύλαξης βεβαίως. Όπως ανέφερε η κυρία Βερχέν, κυρίως πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τους νέους. Η πράσινη βίβλος μας βοηθά να εντοπίσουμε προκλήσεις. Για τον οπτικοστικό τομέα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η διαδικασία. Να είναι ανοιχτό το πνεύμα μας να μην είμαστε συγκεκριμένοι για κάποιο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη διάταξη ε, και να μην πνίξουμε την καινοτομία. Μην χρησιμοποιήσουμε υπερβολικά μέσα για να βρούμε λύσεις. Χρειάζεται αναλογική προσέγγιση. Χρειάζεται ευφυής ε, νομοθεσία και δεν χρειάζεται υπερβολική ρύθμιση. Δεν θέλουμε να πνίξουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη του τομέα. Χρειαζόμαστε την καινοτομία και θα πρέπει να αφήσουμε να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Καναρβέρ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Σαμπίνα και για την παρουσίαση. Της εκθέσεως για την πράσινη βιβλίο. δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ή διαφωνία μεταξύ μας οτιδήποτε και να πούμε τα μέσα μας και είναι ένα διαφορετικό προϊόν, πολιτιστικό προϊόν βέβαια και συστατικό τμήμα των δημοκρατιών μας λόγω της πολυμορφίας που μπορούν να προσφέρουν ή να μην προσφέρουν. Έτσι λοιπόν, οι τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη φυσικά και ως εκ τούτου διαπιστώνουμε ότι το νομικό πλέγμα που έχουμε δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Από την ακρόαση, η οποία νομίζω με πολύ περιγραφικό τρόπο μας έδωσε την εικόνα της κατάστασης, είχαμε δημόσιες, ε, ε, δημόσιες ε, σταθμούς, ιδιωτικούς σταθμούς, παρόχους υπηρεσιών του ε, διαδικτύου ε, και τόσους άλλους που μίλησαν με τοποθετήσεις τελείως αντίθετες ο ένας με τον άλλον, τόσο που σκεφτόμουν εάν κάτι είναι καλό για τον έναν μοιραία θα είναι κακό για τον άλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η δημοσιογραφική ποιότητα, δημοσιογραφική πολυμορφία, όλα αυτά τα θέματα της ελεύθερης ε, έκφρασης και ενημέρωσης που μας ενδιαφέρουν μέσα εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, πρέπει να τα εξασφαλίσουμε, πρέπει να τα εγγυηθούμε χωρίς να ε, προξενήσουμε νέες τρευλώσεις ανταγωνισμού και ώστε να μπορέσει να απελευθερώσει το δυναμικό, το δυναμικό του αυτός ο κλάδος ως οικονομικός κλάδος και να φέρει αποτελέσματα. Τώρα είναι καλή ιδέα αυτή τη πράσινη βίβλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί με την πράσινη βίβλο, με την δική μου έκθεση που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον στη βάση του έχουν απαντηθεί. Όχι σε λεπτομέρειε, αλλά στη βάση του. Πάνω σε αυτό νομίζω μπορούμε να στηριχθούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φεύγουμε τον τροχό και πάλι. Με Εντυπωσιάζει πάντως και κάπως με ενοχλεί θα πρέπει να πω το γεγονός ότι στην Πράσινη Βίβλο ε, προτείνονται και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική για τις συχνότητες, ενώ ε, μόλις ένα χρόνο αφού ετέθη το ζήτημα και χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις σε ερωτήματα, πάνω από 200 τοποθετήσεις είχαμε, πριν λοιπόν δοθούν κάνει απαντήσεις, ε, η Επιτροπή έρχεται με μια πρόταση κανονισμού για την εσωτερική αγορά στις τηλεπικοινωνίες με, τις οποίες, με την οποία μάλλον πρόταση κανονισμού κλείνει το θέμα των συχνοτήτων στις τηλεπικοινωνίες. Ερωτώ λοιπόν τι να την κάνουμε την διαβούλευση, τι να κάνουμε την πράσινη βίβλο, τι να κάνουμε όλα τα ερωτήματα που διατύπονται όταν η Επιτροπή έχει βρει ήδη τις απαντήσεις μόνη της. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν πάει καλά. Για δε την ουδετερότητα του δικτύου που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσουμε στο θεμελιώδες ερώτημα τι είδους πληροφορία, τι είδους εκπομπή θέλουμε να περνάει από το δίκτυο. Και μετά θα μιλήσουμε για την ουδετερότητα του δικτύου. Πρώτα θα κρίνουμε το περιεχόμενο, θα πούμε θα είναι ανεξαρτήτως της προελεύσεως του αντικειμένου της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της πολυμορφίας που θέλουμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και εδώ έρχεται η Επιτροπή με την πρόταση του κανονισμού να κλείσει το θέμα δίνοντας μια πολύ σαφή απάντηση η οποία ξεπερνάει νομίζω τα όρια του κλασικού διαδικτύου και θα απαντήσω δεν θέλω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θέλουμε στην Ευρώπη κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί την ελευθερία της έκφρασης, την πολιτιστική πολυμορφία, την πολυμορφία στην ενημέρωση. Το άλλο θέμα βέβαια, η διαρρύθμιση των πλατφορμών, το τι μπορεί να μπει πάνω σε μια πλατφόρμα και τι μπορώ να βρω κάνοντας, ε, έχοντας την πρόσβαση σε μια πλατφόρμα, σε αυτό θα συμφωνήσω με τη Σαμπίνε, η ρύθμιση της πλατφόρμας θα πρέπει και πάλι να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, να κοιτάξουμε τι νόημα έχει μια πλατφόρμα, ε, ποιος είναι ο ορισμός της. Είναι η Apple, είναι το, η οθόνη σε μια connected, μιας connected TV, μια συνδεδεμένης ε, τηλεοπτικής συσκευής. Ε, όλα αυτά τι είναι. Και νομίζω ότι είναι όλα πολύ σημαντικά και καθοριστική σημασία και πρέπει να μα απασχολήσουν. Αλλά ιδιαίτερα θέλω να πω, να εκφράσω την δυσφορία μου, γιατί ατυπώνονται ερωτήματα από τη μια και από την άλλη, μια άλλη υπηρεσία τη Επιτροπή, προφανώ με ομοφωνία βέβαια μέσα στην Επιτροπή, κλείνει το θέμα, λαμβάνοντα τι αποφάσει για πρόταση συγκεκριμένου κανονισμού. Και διερωτώ με αν αυτό είναι όντω και επί τη ουσία αυτό το οποίο θέλουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αφού δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Έτσι. Διαβάζω εδώ. Η κυρία Νόση, η κυρία Ιμάτ, θα έπρεπε να είναι εδώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Η κυρία Αλόνσο δεν, να δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα. Ονομάζομαι Μάλκοτ και εργάζομαι στην ίδια, ε, στο ίδιο τμήμα. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύγκληση του οπτικοακουστικού τομέα και ήδη αναφέραμε πως υπάρχει, αναφέρθηκε μάλλον πως υπάρχει πράσινο βιβλίο και ότι η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Λάβαμε πάνω από 200 απαντήσεις για αυτή τη διαβούλευση που και αρχίσαμε να τις δημοσιεύουμε και στο ιστότοπό μας. Θα πρέπει να πω πως είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, γιατί έχουμε δημοσιεύσει μόνο αυτές τις απαντήσεις όπου έχουμε τη συμφωνία του απαντώντος να, για δημοσίευση και κάποιες φορές οι απαντήσεις αυτές έρχονται καθυστερημένα. Οπότε πρόκειται για μια εργασία που βρίσκεται σε πρόοδο απίτησαν διάφοροι φορείς, δηλαδή ε, τηλεοπτικά κανάλια, παραγωγή ταινιών, διανομής ταινιών, αλλά και συγκεκριμένοι ε, φορείς που προ... για την προστασία των παιδιών ή για την πρόσβαση, κατασκευαστές του ψηφιακού τομέα. Εχθές έγινε, έγινε μια ανακρόαση που ήταν παρόντες και εκπρόσωποι του τομέα τύπου και βιβλίου. Αυτή τη φορά δεν λάβαμε πολλές απαντήσεις ε, από μεμονωμένα άτομα, αντίθετα με παλιότερες ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που κάναμε νωρίτερα φέτος και ιδιαίτερα ε, μιλήσαμε για ένα ευρύ πεδίο, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πράσινο βιβλίο, ενώ προσπαθήσαμε να μην υπάρχει επικάλυψη με άλλους τομεί. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια στο πράσινο βιβλίο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη αναθεώρησης τη οδηγίας ε, περί υπηρεσιών ε, media. Αυτό μάλλον δεν θα συμβεί κατά διάρκεια αυτή τη θητεία. και δεδομένου του όγκου και της, ε, του πολύπλοκου χαρακτήρα των απαντήσεων που λάβαμε, αναμένουμε πως η ανάλυση θα μας πάρει κάποιο χρόνο και θα χρειαστεί δράση για να σκεφτούμε και να μελετήσουμε τις απαντήσεις. Μέσα σε αυτή την περίοδο προβληματισμού θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, προσδοκούμε την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζοντα το μέλλον τη οπτικοκουστική πολιτική, είτε πρόκειται για νομοθετική δράση είτε για άλλα μέτρα, με στόχο να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη και τι ευρωπαϊκέ αξίε. Σα ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο για τα συμπεράσματα στην κυρία Βερχέιεν. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ του ε, συναδέλφου ε, για τι παρατηρήσει που ετυπώθηκαν σήμερα. Νομίζω ότι επικρατεί ευρεία συνένεση σε πολλούς τομείς. Μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να γίνει πιο σαφής εικόνα για τα πολιτιστικά αγαθά στην Ευρώπη και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις διευκρινήσεις. Ένα θέμα που έθεξε ε, Κάμερ έβερτ. Ε, νομοθετήματα που ήδη είναι ενισχύ και που μπορεί να επηρεάσουν αυτό το οποίο εμείς εδώ προσπαθούμε τώρα σε μια αρκετά πρώιμη φάση να συζητήσουμε. Ναι, υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία είναι ενισχύ σε άλλους τομείς και αυτό το αναφέρω ρητά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, την πολιτική, στην πολιτική για, τα, για τις ε, ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα λοιπά. Ε, και αυτά, όπως είπα, έχουν τεράστιες επιπτώσεις στον χώρο των οπτικοακουστικών, στον τομέα της σύγκλησης που μας ενδιαφέρει στο σημερινό κόσμο ιδιαίτερα. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, πιάσαμε το ε, θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε από πλευράς των, της λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης». Δεν μπορούμε να αποκόψουμε ένα άλλο θέμα, ε, από το, ένα θέμα από το λοιπό πλέγμα σχέσεων ε, στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού. Επομένως, αντιλαμβάνομαι τη δυσφορία που αισθάνεται η συνάδελφος Κάμερ Εβερτ. Πολλά πράγματα έχουν γίνει ίσως μερικός, όχι επαρκώς ε, στον χώρο αυτόν, αλλά ίσως η απάντηση δεν είναι να τα απορρίψουμε σε λίβδιν. Θα πρέπει να μελετήσουμε τι είδου επιπτώσεις μπορεί να έχει το κάθε νομοθέτημα σε αυτά που έχουμε εμείς κάνει και κυρίως μακροπρόθεσμα για να μπορέσουμε να λάβουμε τις απαντήσεις. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι περίτη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και μπορούμε και τώρα και με την πρόταση μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες ακόμη να κάνουμε τη γενική αυτή συζήτηση και να επισημάνουμε τα σημεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αντίστοιχα και με ιδέες και προτάσεις που προκύπτουν από την πράσινη βίβλο. Άλλωστε το είδαμε και στην τελευταία ολομέλεια ότι αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί στην ε, Επιτροπή με μεγάλη δυσκολία δεν, ε, θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην συμβεί αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν, δηλαδή αποφάσεις που έχουμε λάβει με μεγάλη δυσκολία εδώ στην Επιτροπή, με μία και μόνη ε, ψήφο και πολύ εύκολα να ανατρέπονται και να καταργούνται από την Ολομέλη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και βέβαια με μεγάλη χαρά περιμένω τη συνεργασία για την έκθεση που θα ακολουθήσει αυτή την ε, πράσινη βίβλο. Σας ευχαριστώ. Οπότε περνάμε στο τελευταίο, στα ένατο και τελευταίο σημείο της σημερινής συνδέδεξης, για το οποίο θα ακούσουμε την παρουσίαση των νικητών του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνος το 2013. Το βραβείο αυτό ξεκίνησε από το 2008 ως κοινή πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Μάγνος με στόχο να βραβεύει προγράμματα που έχουν υλοποιήσει νέοι Ευρωπαίοι ανάμεσα στα 16 και τα 30 έτη ηλικίες για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ε, ολοκλήρωση ανάμεσα στους νέους. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας επιλογής ε, ε, έχουν σε δύο στάδια. Κάθε πρόγραμμα έχει εγκριθεί από ένα εθνικό όργανο και από ένα διεθνές όργανο στο οποίο συμμετέχουν και δύο ευρωβουλευτέ. Στο... Έπειτα έρχονται στην Κεντρική Επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο Σούλτ, δύο ακόμα ευρωβουλευτέ και τέσσερι εκπροσώπου του Ιδρύματο Καλομάγνο. Και έτσι η Κεντρική αυτή Επιτροπή επιλέγει τα τρία καλύτερα προγράμματα. Και όλοι οι εθνικοί νικητέ ε, συγκεντρώθηκαν ε, πριν από, τρεις, πριν από ένα μήνα στον Κουσγκράνα. Το πρώτο βραβείο δόθηκε στο σχέδιο τη Λετωνία, ε, το σχέδιο της ζωής μου για την πρόθεση της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης ανάμεσα στις γενναίες. Νέοι από διάφορες χώρες, ε, με ηλικιωμένους από διάφορες ε, χώρες συγκεντρώθηκαν στη Λετωνία. Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν ο στόχος της Ευρώπης από την Πολωνία που ήταν επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών από φοιτητές που προέρχονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το πρώτο δε βραβείο το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνου δόθηκε στην Ευρώπη στο, στην ε, μέλλον. Βλέπει πώς, ε, το πρόγραμμα αυτό πώς με βίντεο ε, φωτογραφίες και blog πώς οι νέοι βλέπουν το μέλλον τους στην Ευρώπη. Και σήμερα καλωσορίζουμε εδώ τους τρεις ε, νέους από τις συνοικήτριες ομάδες. Εστονία, η ιστορία της ζωής μου, η κυρία Καλντόγια, είναι εδώ. Ναι, χρειάζεται και το χειροκρότημα. La seconda classificata dalla Polonia η δεύτερη νικήτρια από την Πολωνία είναι η κυρία Σενίκα. Ελπίζω να το, ε, να το πρόφερα καλά. Και η νικητές, γιατί είναι, μια, είναι ένα ζευγάρι, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Η κυρία Ρόποντρα και ο κύριος Λουίς Βαλδαράδο Μαρτίνες και η κυρία Βένερα. Συγχαρητήρια. Allora daremo la parola ora. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μαρτίνες και στην κυρία Ρένερ για πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό που έφτιαξαν και να καταλάβουμε πώς λειτουργήσαν. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό που μια φορά ε, αφιερώνετε λίγο χρόνο να ακούσετε τους νέους. Το πρόγραμμα ε, είναι μια συνεργασία που κάνουμε το Ιντερέλ και δίνουμε τη δυνατότητα σε πρέσβεις να ταξιδεύουν στην Ευρώπη για ένα μήνα, ε, παίρνοντας συνεντεύξεις από τους τους νέους στην Ευρώπη, τι θέλουν από την Ευρώπη μέχρι το 2020. Επιχειρηματικότητα των νέων, βιωσιμότητα, συμμετοχή των νέων. Για ένα μήνα δηλαδή συγκεντρώναμε τις απόψεις των νέων από όλα τα κρατημέλη και μάλιστα ήταν αρκετά αυστηρή για την κατάσταση της Ευρώπης. Την επέκριναν Πολύ καλές συστάσεις έκαναν για τα θέματα που κανονικά ε, δεν ακούγονται μέσα στα θεσμικά όργανα. Θέλαμε να δώσουμε ένα φρέσκο, ένα ζωντανό και θετικό μήνυμα για την Ευρώπη από τη νέα γενιά που καταλαβαίνει ότι το να μην υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επιλογή. Για εμά η Ευρώπη είναι καθημερινή πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε τα ωφέλη και τι ευκαιρίε που προσφέρει η Ευρώπη, αλλά στι πόλει, σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτε δεν καταλαβαίνουν πάντοτε και ήταν αρκετά αυστηροί. Είναι δική σας δουλειά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές οι πρωτοβουλίες ε, και, ε, όχι, και οι καλές αποφάσεις που λαμβάνετε εδώ να φτάνουν και στους πολίτες. Μια πολύ συχνή παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη παιδείας και κατανόησης για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι, ποιος είναι ο αντίκτυπός του στην καθημερινή ζωή. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί θέλω και οι συνάδελφοι να εκφραστούν, αλλά ίσως ε, να σας παραθέσω ένα αίτημα, ειδικά πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ, ήταν ότι αν θέλουμε να αλλάξει αυτό που κάνει η Ευρώπη και θέλουμε συμμετοχή των νέων, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε στοχευμένες εκστρατείες και να εξηγούμε στους νέους ποια είναι τα εφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την Ευρώπη, αλλά κυρίως να υπάρξουν νέοι εδώ σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Οι νέοι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούνται ότι προσωπεύονται εδώ και γι' αυτό είναι καθήκον των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ομάδων να εξασφαλίσουν προκαλέσουν περισσότερη ε, παρουσία νέων, ώστε οι νέοι να θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ε, και να ενημερωθούν για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχετε πολύ, πολύ δουλειά εδώ και δεν τα καταφέρνετε και πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται για τους νέους. Οι νέοι περιμένουν πολλά από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρένα, θέλει να πει κάτι. Α, όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Και περνάμε στην δεύτερη νικήτρια, την κυρία Σινίκα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Κατερίνα Σινίσκη και είμαι η συντονίστρια αυτού του προγράμματος και έχω τη χαρά και τη τιμή να σας παρουσιάσω το πρόγραμμά μας που είναι μια Ευρω... ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Ανακαλύπτε την Ευρώπη». Ήθελα να σας πω τι είναι ακριβώς αυτή η ένωση το Erasmus Network. Δημιουργήθηκε το 87, το 1987 ως ένας ε, σύνδεσμος για τη στήριξη του προγράμματος Erasmus. Τη διεθνή δηλαδή ανταλλαγή φοιτητών. Θέλαμε να βοηθήσουμε δηλαδή τους ε, φοιτητές ε, αλλά και να ε, ε, τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν την κουλτούρα μας στην Πολωνία. Γι' αυτό και ερχόμαστε σε επαφή με τους φοιτητές ε, του Εράσμου που έρχονται στη χώρα μας. Κάνουμε μια μεγάλη σειρά από προγράμματα ε, που καλύπτουν ένα μεγάλο πεδίο και γι' αυτό θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τρία-τέσσερα προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από το δικό μας ε, τμήμα στην Πολωνία. Υπάρχει το κοινωνικό Έρασμος που θέλει να καλέσει τους φοιτητές που συμμετέχουν στο Εράσμο στην Πολωνία ώστε να μπορέσουν να αναμειχθούν με την τοπική κοινότητα. Τους ε, κάνουμε να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, ένα είδος μιας μικρής Ολυμπιάδας. Το άλλο πρόγραμμα λέγεται «Ανταλλαγή ε, δεξιοτήτων να δείξουμε ποιε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ε, αναπηρίες. Να μιλήσω λίγο και για την ιστορία. Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε το 2003 μετά από πρωτοβουλία των φοιτητών της ε, Εμπορικής Σχολής ε, της Βαρσοβίας και στρέφεται και στους ξένους, όχι μόνο στους Πολωνούς. Το 2008 η Ένωσή μας αυξήθηκε περισσότερο γιατί δόθηκε ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές Πολωνίας να συμμετέχουν. Καλύπτουμε δηλαδή την Εθνική Επικράτεια και το 2009 ευρωπαϊκό χαρακτήρα απέκτησε αυτό το πρόγραμμα που θέλει στην ουσία να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στους Πολωνούς και τους Ευρωπαίους φοιτητές. Θέλουμε να δείξουμε την πολυμορφία της Ευρώπης μέσω όπως σας είπα, με εκθέσεων φωτογραφίας, διαχωνισμών. Έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Φέτος προσθέθηκε και μία τέταρτη. Η κατηγορία της, ε, των φίλων, των ταινιών. Έχουμε τοπικό επίπεδο στην Ένωσή μας, είναι υπεύθυνη για την πρόθεση στα σχολεία, είναι πολύ σημαντικό διάβλος επικοινωνίας γιατί έτσι φτάνουμε στους αποδέκτες μας πιο εύκολα, έπειτα έχουμε περιφερειακό επίπεδο και εκεί γίνεται ενημέρωση σε περιφερειακό επίπεδο γιατί έτσι εκεί σε αυτό το επίπεδο συλλέγουμε τις φωτογραφίες, ε, συλλέγουμε το 10% και μετά περνάμε στο ε, κεντρικό επίπεδο όπου συντονίζονται, όλες οι λειτουργίες για την απόκτηση ε, ε, κονδυλίων, για την ανέβρεση κονδυλίων, για την ε, διοργάνωση εκθέσεων, για την αναζήτηση εταίρων και έπειτα γίνεται στο τέλος μια τελική εκδήλωση όπου ε, ε, ανακοινώνεται ο νικητής. Είχαμε μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε πολλούς εταίρους και εργοδότες ανάμεσα σε τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Σούμαν, γιατί μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε ένα καλό ε, βραβείο για τους νικητές. Ε, επίτα να σας πω ότι διοργανώσαμε ε, και μια κινητή έκθεση και σε μια τελευταία εκδήλωση καλέσαμε όλους τους νικητές και την Κρητική Επιτροπή καθώς και πολλούς θεατές. Δύο δε ραδιοφωνικές εκπομπές αφιερώθηκαν σε, αυτό, σε αυτές τις εκδηλώσεις. στις προηγούμενες εκδοχές οι φωτογραφίες ήταν γύρω στις 3.000 που είχαμε συλλέξει, ενώ φέτος μπορέσαμε να φτάσουμε σε πολύ περισσότερους ε, συμμετέχοντες και φτάσαμε στις 3.800 φωτογραφίες. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ ενδιαφέροντα από για μας τους φοιτητέ, ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέροντα για εσάς τους πολιτικούς, αλλά έτσι εμείς μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες ένταξης, marketing, δουλεύουμε σε ομάδες, ε, ε, μπορούμε να αναπτύξουμε και τις ε, ηγετικές μας ικανότητες, αν έχουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά λοιπόν στην Πολωνία, γιατί έτσι αποκτούμε εμπειρίες και που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αργότερα στον χώρο της εργασίας, αν βρούμε Σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μας. Και τώρα το λόγο έχει... Ε, Καλδόγια, πρέγω. Η κυρία Καλδόγια. Hello from my side also and thank you for having us. Γεια σας. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Όπως είπε και ο Μαρτίνες, οι νέοι δεν μπορώ να μιλάνε συχνά σε τέτοιους χώρους. Είμαι θα ευγνωμονε για τη δυνατότητα που μας δίνεται. Και όπως θα ακούσατε, στην Εστονία θέλαμε να συναθήσουμε διάφορες γενιές. Ηλικία 15 με 25 και μετά 60 με 70. Η ιδέα διεθνής ανταλλαγή νέων κάτι κοινό στην Ευρώπη. Επιπλέον όμως φέραμε μαζί και 10-15 ηλικιωμένους από την Εστονία ανάμεσα στα 60 και 70. Κάναμε τα πάντα μαζί για δύο εβδομάδες. Θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι όλοι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, δεν πρέπει να υπάρχουν στερεότυπα περί και νέων, Εδώ είναι, δεν υπάρχουν πολλοί νέοι στο κοινοβούλιο που θεσπίζουν νομοθεσία, δεν ακούγεται η φωνή των νέων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη συχνά τις ανάγκες των νέων. Θέλαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν διάλογο με αυτή την προσπάθεια. Θα έλεγα ότι ήταν επιτυχές το πρόγραμμα, καλυφθήκαμε πολύ από τα ΜΜΕ και στην Εστονία και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Πορτογαλία κλπ. Έληξε για φέτος το πρόγραμμα και στον οργανισμό μας επιλέγουμε κάθε χρόνο ε, νέα θέματα. Δυστυχώς έληξε αυτή η προσπάθεια. Ίσως θα μπορούσαμε να πνεύσουμε και άλλες χώρες να κάνουν κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μακλάρκιν ζήτησε το λόγο. Σας καλωσορίζω όλους. Είναι υπέροχο το ότι μειώνεται το μεσόωρο ηλικία στην αίθουσα. Εγώ είμαι νεότερη, το νεότερο μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι 35 ετών όμως. Και είσαστε πολύ νεότεροι ακόμα και από μένα. Είναι πολύ σημαντικό που εμείς στο Κοινοβούλιο ακούμε τους νέους και προσπαθώ να εκπροσωπώ τις απόψεις σας στο μέτρο του δυνατού. Το κάνουμε σε αυτή την Επιτροπή επίσης, ανεξάρτητα ηλικίας είναι η Επιτροπή, η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, είναι και η Επιτροπή Νεολαίας που προσωπούμε τις απόψεις των νέων, προσπαθούμε τουλάχιστον και συζητάμε θέματα που είναι σημαντικά για σας. Και προσπαθούμε να θυμόμαστε πώς είναι να είναι κανείς νέος συνεχώς όταν συζητούμε. Είναι πιο δύσκολο για μερικούς από ό,τι για άλλους. Τα προγράμματά σας είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μα μου τόσο έξυπνοι όταν ήμουν στην ηλικία σας να σκεφτώ ε, να, να τέτοια προγράμματα όπως αυτά που αναφέρατε ταξιδεύοντας με το τρένο και τι εικόνες θα μαζέψατε και απόψεις. Θα, θα με ενδιαφέρε να ακούσω τι απόψεις μαζέψατε από το, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες από γενιά σε γενιά, ανταλλαγή μεταξύ γενιών. Να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των γενεών, να καταλαβαίνουμε τους δε, να μην λένε οι μεν εμείς καταλαβαίνουμε τον καινούριο κόσμο και εμείς καταλαβαίνουμε τον παλιό κόσμο. Και σαν φωτογράφος, μανιώδης, και εγώ θα ήθελα να δω τις φωτογραφίες. Και είδα πόσους υποψηφίους είχατε για τους... Ε, ε Πώ υποψηφιώτε, 3.600 φωτογραφίε. Εγώ είχα οργανώσει στην εκλογική μου περιφέρεια μια τέτοια αγωνισμό και είχα λιγότερο από 100 φωτογραφίες. Άρα είσαστε πολύ πιο δημοφιλείς ή καλύτεροι στην επικοινωνία από ότι είμαι ακόμα και εγώ που είμαι πολιτικός. Πολύ καλά τα κάνετε παιδιά, τα καταφέρατε. Μπράβο. Χρησιμοποίησατε το έρασμο που είναι από τα θετικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το προωθήσατε και δείξατε ότι χρειάζεται διαπολιτισμικό διάλογο για να εκτιμηθούν οι διάφορε κουλτούρε που υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στα διάφορα κράτη-μέλη και στο κοινοβουλίο. Ευχαριστώ που ήρθατε και μα θυμήσατε να μην σα ξεχάσουμε στι ευρωεκλογέ. Κυρία Βερέν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε και για τα προγράμματα που ετοιμάσατε. Και στο Άχελ, τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, μας ε, ενδιαφέρουν πάρα πολύ και πρέπει να πω ότι με συναρπάζει ο ενθουσιασμός που δείχνετε εσείς για την Ευρώπη. Αυτό είναι και το κοινό, νομίζω, χαρακτηριστικό όλων σας των προσπαθειών και επίσης νομίζω ότι εσείς μπορείτε να δείξετε, να, δω, να μεταδώσετε στους πολίτες τι σημαίνει το πνεύμα, το ευρωπαϊκό πνεύμα. Σε ένα μόνο θα ήθελα να φέρω αντίρρηση. Έχουμε, σε σχέση με άλλα κοινοβούλια εθνικά, πολύ μεγάλο ποσοστό νέων. Δεν έχουμε μόνο την κυρία Μακλάρκινγκ που είναι αρκετά νέα, αλλά αν κοιτάξετε και τους βοηθούς μας, τους συνεργάτες μας εδώ στο κοινοβούλιο, θα δείτε ότι είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι με τη δραστηριότητά τους, με τρόπο δραστήριο, ε, συνδιαμορφώνουν την πολιτική στην Ευρώπη. Μην ε, μας λέτε λοιπόν ότι στέλνουμε τους ε, παππούδες και τις μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως παλιότερα συνέβαινε. Έχουμε ένα νεαρό κοινοβούλιο συγκριτικά, ένα ζωντανό και ζωτικό κοινοβούλιο και νομίζω ότι Βλέπετε κι εσείς από τη σημερινή σας εμπειρία ότι δεν συνομιλείτε μόνο για, με και παππούδες. Νομίζω όμως ότι πρέπει να επιμένουμε ιδιαίτερα στην ε, εμπλοκή των νέων στην ε, συζήτηση αυτή. Χρειάζεται μια νέα αντίληψη για το μέλλον έχω πολλές φορές έχω την ευκαιρία να συζητήσω με νέους από διάφορες γενναίες για πράγματα τα οποία ίσως για τον πιο ηλικιωμένο είναι αυτονόητα ε, για τον οποίο μάλλον είναι αυτονόητα αυτά τα οποία ο πιο ηλικιωμένο δεν έχει ζήσει. Δεν θεωρεί τόσο αυτονόητα. Δηλαδή αυτό που έχει γνωρίσει τον πόλεμο, την, ε, το σπαραγμό, την πείνα, την, ε, τη δικτατορία. Για εσά μπορεί η δημοκρατία και η να είναι κάτι το αυτονόητο. Εσείς με, με τεράστια ευκολία πήγατε από το ένα κράτο στο άλλο για να σπουδάσετε με τι ανταλλαγέ Εράσμου. Υπάρχουν πράγματα, είναι όλα αυτά όμω πράγματα τα οποία δεν ήταν δεδομένα για τι προηγούμενε γενιέ, τα οποία εσεί έχετε εγγυημένα και τα οποία πρέπει να διαφυλάξετε και με την κοσμοθεωρία σας. Αυτό ε, που θέλω δηλαδή να πω είναι ότι φορείς των ε, ιδεοδών των αξιών της Ευρώπης θα είναι οι νέοι, οι νέοι εκείνοι οι οποίοι θα στρατευτούν και που θα παρουσιάσουν έργο και σχέδιο και όραμα για την Ευρώπη, για τη συνεργασία. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, γιατί με τα σχέδιά σας έχετε υλοποιήσει αυτήν, ε, την, αυτό μας το όραμα ε, σας χρειαζόμαστε. Σας χρειαζόμαστε ως πρέσβης, ως φορείς αυτού του μηνύματος το οποίο θα πάει και στους άλλους νέους, τους νέους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό χωρίς ίσως και να κερδίσουν, τους νέους που μπορεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, σε κάποια άλλη ευκαιρία να συναντήσετε μέσα από τα κομμένιους ή τα εράσμους, ε, που δεν είχαμε πάντα την ευκαιρία εμείς να δούμε, αλλά πάνω απ' όλα με μια υποδειγματική υποστήριξη αυτού του οράματος που είναι η Ευρώπη. Και νομίζουμε ότι έτσι μπορεί να φτάσει αυτό το μήνυμα σε όλους τους νέους που δεν δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρώπη σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη στράτευση και τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι υπόθηκαν τα πάντα, αλλά και εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για μια απίστευτη στράτευση και αγώνα που δεν είναι καθόλου αυτονόητο στην Ευρώπη, στον οποίο έχετε αποδειχθεί. Ε, ιδιαίτερα δε Αισθάνομαι υπερήφανη γιατί είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην Εθνική Εφορευτική Επιτροπή από τη Γερμανία που μου επέτρεψε με αυτόν τον τρόπο να έρθω πιο κοντά στο εγχείρημα, κοιτάζοντα όλε τι προτινόμενε ιδέε και να δω πόσο τεράστιο πλούτο και ποιότητα ε, ιδεών και σχεδίων ε, προτάθηκε από τους νέους της Ευρώπης. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να διαμορφώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η Σαμπίνα είπε ότι πολλά πράγματα για σας είναι αυτονόητα. Μιλάμε για κρίσεις, μιλάμε για οικονομικά, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ποια είναι η καρδιά της Ευρώπης και τέτοιου είδους ε, σχέδια πιστεύω μπορούν ιδιαίτερως να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής, στην προαγωγή λίγο ακόμα αυτής της ευρωπαϊκής ταυτότητας και νομίζω μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε κάποιες τάσεις εθνικιστικές ή ακροδεξιές, λαϊκιστικές που βλέπουμε να αναφύονται σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Εσείς είστε η γενεά εκείνη η οποία θα πρέπει να διευρύνει ακόμη αυτή την Ευρώπη μέσα στην οποία ζούμε. Θα έχετε εσείς το καθήκον αυτό και με τις ευκαιρίες που σας δίνουν τα προγράμματα ανταλλαγών, εράσμους και άλλα, που γνωρίζετε ε, νέους από άλλες χώρες, που ταξιδεύετε, που συμμετέχετε σε ε, συνεργασίες ακόμη και θεατρικές και ούτω καθεξής, μπορείτε να αποτελέσετε τον κρίκο. Τον κρίκο αυτό που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει η Ευρώπη και που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας παρακαλώ να μην εγκαταλείψτε τον αγώνα. Αυτή την δημιουργικότητα, αυτή την αποφασιστικότητα τη χρειάζεται η Ευρώπη. Και θέλουμε αυτό το σχέδιο για την ειρήνη να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες, αν δεν κάνω λάθος, ζητούσε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο σχόλιο από την πλευρά μου. Μεγάλη πρωτοβουλία για μας τους νέους να έρθουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή για να παρουσιάσουμε τα θέματά μας, αλλά και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αρκετά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου λοιπόν. Θα έπρεπε η Επιτροπή να δει πόση σημασία δίνουμε στις φωνές των νέων, παρά το γεγονός ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά στον αφορά τα προγράμματα για τι διαπραγματεύσει και του προπολογισμού. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά όταν οι νέοι έρχονται σε αυτό το θεσμικό όργανο, πώ αισθάνονται στο σπίτι του, όταν εμεί η νεότερη γενιά που βλέπουμε την Ευρώπη σαν κάτι που πρέπει να υπάρχει και είμαστε η γενιά που ζήσαμε με την Ευρώπη καθημερινά και δεν μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη, μια, τη ζωή χωρίς Ευρώπη, επιστρέφουμε στη, χώρα μας και μας χτυπάνε οι, οι γονείς και οι παππούδες λένε δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη πια. Και ερχόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τη βοήθεια που είμαστε στην Ευρώπη και εσείς απουσιάζετε, Ίσως θα έπρεπε κάπως αυτό να το κρίνετε. Πού είναι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποστηρίζουν του νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να σας πω ότι όντας ο νεότερος σε αυτή την επιτροπή όπως μπορείτε να δείτε γέρασα προήμως διότι η πολιτική στην Ευρώπη καμιά φορά δημιουργεί πάρα πολλές ανησυχίες. Φαίνονται πιο ηλικιωμένο τώρα πια στην επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και λυπάμαι και το λέω ονόματι της ε, Προέδρου που υπάρχουν πολύ λίγοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Προφανώς είναι κάτι που θα το πούμε στους συναδέλφους, ότι βλέποντας τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες ε, που ανελήφθησαν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Όμως ευχαριστούμε τους συναδέλφους που όμως παρέμειναν εδώ και ήταν παρόντες και σας άκουσαν. Σας ευχαριστώ. Πέρα στη συνεδρία σας θα παραμείνουμε εδώ για τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όποιος είναι συντονιστή σας μείνει και κλεισμένο το θηρόν θα γίνει η συνεδρίαση. Παρακαλώ οι υπόλοιποι αν έχουν την καλοσύνη να αποχωρήσουν.